ένσταση, τότε ε, ο ορισμός αυτών των μελών θεωρείται εγκεκριμένος. Ο κύριος Ντάνιελ Φαντεστούπ με, μου έχει πει ότι παρετείται ως Ευρωβουλευτής ε, και ε, αναδράμει αυτή η παρέτηση στην, ανατρέχει μάλλον συγγνώμη την πρώτη του 2011 Σήμερα με το άρθρο 4 παραγράφη 1 3 του κανονισμού το κοινοβούλιο επιβεβαιώνει το ότι χειρεύει η θέση του και θα ανατρέχει ακριβώς αυτή η χειρία σε εκείνη ημερομηνία. Επίσης, οι Ολλανδικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι έχει οριστεί την κατάσταση του, του κύριου Ντάνιελ Φαντερστούπ από τον κύριο Άουγκε Ζέλστρα. Και η κατάσταση θα υπολογίζει ότι λαμβάνει χώρα από 13 Σενάτου 2011. Παρίστατε εδώ ο νέος συνάδελφος. Είστε εδώ. You Καλώς ορίσατε. Właściwe organy szwedzkie poinformowały mnie o zastąpieniu Επίσης, οι αρμόδιες σουηδικές αρχές μας ενημέρωσαν σε σχέση με την αντικατάσταση της κυρίας Εύα Μπριτ Σβένσον. Αντικατάστατης είναι ο κύριος Μίκαελ Γκούσταυσον και ε, θεωρείται ότι ισχύει αντικατάσταση από τις 22 Ιανουαρίου του 2011. Παρίσταστε εδώ, συνάδελφε. Όχι, δεν παρίσταται ο συνάδελφος Γκούσταυσον. Επίσης, ε, πάλι καλωσόρισαν όρισαν ε, οι νέοι συνάδελφοι, τους καλωσορίζω εκ μέρους όλου του σώματος και σας ε, υπενθυμίζω ότι δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού μας μέχρι ότου έχει γίνει παλήθευση του διορισμού τους και μέχρι ότου δεν έχει κρυθεί ε, τυχόν ένσταση ε, λαμβάνουν τα, τα έδρανά τους, ε, λαμβάνουν τις θέσεις τους οι συνάδελφοι σε όλα τα όργανα του Κοινοβουλίου, απολάβουν όλων των δικαιωμάτων, ε, όμως θα πρέπει πρώτα να έχουν ε, υπογράψει την ε, δήλωση ότι